πρωινή συνεδρίαση. Η μέσα διάταξη προβλέπει την κοινή συζήτηση σχετικά με τα δραστηριότητε πιστοτικών ενδυμάτων και την εποπτική ε, προληπτική συγγνώμη εποπτεία πιστοτικών ενδυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων ε, του κυρίου Κάρα. Δίνω τον ε, λόγο στον κύριο Κάρας. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, Η έκθεση που έχουμε συζητήσει και κυρίω το αποτέλεσμά τη είναι μεγάλη επιτυχία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεγάλο, ε, μεγάλη επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση ω χρηματοπιστωτική αγορά, μεγάλη επιτυχία για την Ευρώπη ω οικονομικό κέντρο για την εσωτερική αγορά. Και διασώζουμε, ε, ρυθμίζουμε μάλλον όχι κάποιες τράπεζες, αλλά όλες τις τράπεζες ρυθμίζουμε με συνεννόηση και σε συνεννόηση με τους πάντες τη λειτουργία των ε, τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ε, σε συνεργασία το Κοινοβούλιο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της αγορές, και οι 8.200 τράπεζες των ευρωπαϊκών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ε, σταθεροποιηθούν χάρη στις ε, προβλέψεις αυτές. Θα εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση της πραγματικής αγοράς, τη διάθεση πιστώσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα ενισχύσουμε την ε, τον ισότιμο ανταγωνισμό στις, μεταξύ των τραπεζών στην ευρωπαϊκή αγορά. Αποφασίζουμε λοιπόν κυρίες και κύριοι σήμερα διατάξεις οι οποίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο ε, των ρυθμίσεων που έχουμε στο μέλλον να υιοθετήσουμε και αποτελούν την ε, βάση της ε, λειτουργίας από εδώ και μπρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν αυτό το δρόμο, αυτή την επιτυχία, με μια έκθεση πρωτοβουλίας τον Σεπτέμβριο του 2010, διότι μέσω αυτής της έκθεση πρωτοβουλία και τη αντίδραση που επεφύλαξε στο έγγραφο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετέθησαν τα πρώτα ε, τα πρώτα λιθάρια στο δρόμο αυτό που στρώθηκε για την επιτυχία. Και αυτό επειδή το Κοινοβούλιο, ενωμένο πάντοτε, ασχολήθηκε με την ουσία του ζητήματος και δεν προσπάθησε να προβάλλει ε, τις διαφορές. 38 υπέρ καμία ψήφος κατά για την έκθεση πρωτοβουλία. 44 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά για την ε, ψηφοφορία επί της ε, προτάσεως Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καμία κοινοβουλευτική ομάδα δεν διαφοροποιήθηκε. Και εδώ τι έχουμε να, να ε, φέρουμε στις προτάσεις μας. Έχουμε να κάνουμε με την εφαρμογή στην πραγματική αγορά, την μετάθεση στην πραγματική αγορά των συνθήκων ανάπτυξης και λειτουργίας και ταυτόχρονα τη διεύρυνση της ε, εταιρική διακυβέρνησης και στις τράπεζες. Έχουμε περισσότερο λοιπόν κεφάλαιο στη θέση μα, διπλασιάζεται το κεφάλαιο. Ναι, έχουμε δύο νέα ορόσημα ε, ρευστότητα. Ναι, ε, μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο, μπορούμε να αυξήσουμε την. Ε, προστασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους και έχουμε τη δυνατότητα έτσι να προσφέρουμε ισότιμες συνθήκες πρόσβασης με αποκεντρωμένο τομέα, με προσδιορισμό και της πριμοδότησης, ε, των πριμ δηλαδή, που θα αποτελούν ε, ένα πολλαπλάσιο των μισθών, των μηνιαίων μισθών, ε, έχουμε να κάνουμε με την προστασία και των χρημάτων του φορολογουμένου από την φοροδιαφυγή. Έχουμε να κάνουμε με την ε, ε, ενίσχυση των ευθυνών στις ηγετικέ θέσεις των στελεχών με περισσότερη διαφάνεια και ως εκ τούτου με μια βάση για καλύτερη εποπτεία των τραπεζών. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να απευθυνθώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Προεδρία, το ε, σύνολο των συναδέλφων, βουλευτών, τον σύνολο του προσωπικού του Κοινοβουλίου για να ευχαριστήσω για την προσπάθεια στην οποία αποδεθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια ε, και την σαφή απόφαση και απάντηση που δίνουμε στις μεγάλες προκλήσεις ότι θέλουμε ένα σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα, θέλουμε υγιείς και στεναρές τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Υπουργός Κάιτον. Ή Υπουργός, συγγνώμη. Ε, ε, Αγαπητά μέλη, το πακέτο, το νομοθετικό πακέτο αποτελεί, ε, είναι απότοπο, απότοκο, με συγχωρείτε, της ε, στεναρής εργασίας των θεσμικών οργάνων. Και θα ήθελα να τονίσω τη συνεισφορά της Πολωνικής, Δανικής και Κυπριακής Προεδρίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Κάρας, τον ε, εισηγητή, την κυρία Νόλς, την πρόεδρο της ΕΚΟΝ, και τους Bauman, Lambers και Ford. Και Ford γιατί συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Χαίρομαι διότι φτάσαμε σε ένα πολιτικό αποτέλεσμα και αυτό σημαίνει ότι οι νέοι κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν από την 1η Πρώτου του 2014. Το πακέτο αυτό αποτελεί το επίκεντρο του, ε, της ενιαίας αγοράς και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ε, ε, διεθνείς μας δεσμεύσεις σε σχέση με τη Βασιλεία 3 και τις απαιτήσει ρευστότητας θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις για να είναι πιο ανταγωνιστική και να φτάσει σε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό θα πρέπει να εξισορροπήσουμε τα, ε, την ε, αύξηση κεφαλαίου και την ρευστότητα των τραπεζών, ιδιαίτερα σε σχέση με τις παροχές προς τις ΜΜΕ. Νομίζω ότι το πακέτο αυτό ε, δίνει πραγματικούς, ε, πραγματικά κίνητρα για να τα επιτύχουμε. Ενώ οι συμφωνίες της Βασιλείας αφορούν τις μεγαλύτερες παγκόσμιες τράπεζες, εμείς ασχολούμεθα και με τις τράπεζες και με τις επιχειρήσεις, επιχειρήσεις επενδύσεων. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμόρφωσή μας με τους παγκόσμιους κανόνες και με την προληπτική εποπτεία. Γνωρίζετε τα βασικά σημεία του κειμένου το οποίο θα ψηφίσετε σήμερα. Θα ήθελα όμως να τονίσω ορισμένα σημαντικά σημεία. Το πλέον θεμελιώδες είναι ότι οι τράπεζες θα πρέπει να κατέχουν περισσότερο και καλύτερο κεφάλαιο και να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τις προαπαιτήσεις ρευστότητας. Έτσι δεν θα αναλαμβάνουν υπέρμετρο κίνδυνο. Επίσης, πέρα από την αντιμετώπιση του συστημικού κινδύνου, ε, λαμβάνοντας υπόψη ε, συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση συστημικών κινδύνων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι κανόνες και τα, ε, και τα μέτρα ανάσχεσης θα πρέπει να λάβουν υπόψη ε, όλα, όλη την διαδικασία της προληπτικής εποπτείας. Μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε και να ανασχέσουμε τους κινδύνους, τους ε, μακροπροληπτικούς και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων της Βασιλείας και παραβίαση της προληπτικής εποπτείας. Έτσι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη διαδικασία και την αναλογία μόχλευσης και κάλυψης ρευστότητας μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής των απαιτήσεων της Βασιλείας και της προληπτικής εποπτείας καθώς και τον χρηματοπιστωτικό τομέα και την ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τις επιδοτήσεις αναχώρα καθώς και τον ε, τζίρο και τον αριθμό εργαζομένων. Από το 2014 όλα αυτά θα κοινοποιούνται στην Επιτροπή και από το 2015 θα πρέπει να είναι διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία δημοσίως. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την οροφή των πόνους που καταβάλλονται ε, στους υπαλλήλους της τράπεζας και την διαδικασία καταβολής 25% αυτού του μπόνους με συγκεκριμένα ε, μέτρα, με συγκεκριμένες διαδικασίες όπου θα υπάρξουν και χαμηλότερες καταβολές. Ως προς την διαδικασία εποπτείας θα τονίσουμε το ρόλο της ΕΑΤ με βάση του, το ρόλο εποπτείας που έχει αναλάβει. η Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, η συμφωνία μας σε αυτό το νομοθετικό πακέτο δεν σημαίνει ότι έχει λήξει η εργασία αυτή. Θα πρέπει να αποτιμήσουμε την όλη διαδικασία εφαρμογής της νομοθεσίας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας αριθμός ε, ρητρών αναθεώρησης που καλύπτουν την ε, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της οικονομίας το καθεστώς που ισχύει σε ε, μεγάλες εκθέσεις, καθώς και τις απαιτήσει για την κάλυψη της ρευστότητας και την εποπτεία των τραπεζών. Θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αποτελεί καλή έκβαση και ελπίζουμε ότι θα υποστηριχτεί από το Κοινοβούλιο. Αποτελεί ένα βασικό βήμα για την καλύτερη ρύθμιση της βιομηχανίας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και έτσι θα οικοδομήσουμε εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών στον χρηματοοικονομικό τομέα της Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Ο Επίτροπος Μπαρνιέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα σε όλες και όλους. Κύριε Βουλευτέ, σας επέβαλα αυτό το κείμενο τον Ιούλιο του 2011. Σήμερα περνάμε σε μια ε, περαιτέρω φάση θα έλεγα ότι είναι ακροκονία λήθος του Single Roll Book με τις 8.300 ε, τράπεζες ε, που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις σε ποιότητα, ποσότητα των ιδίων κεφαλαίων, ε, νέες απαιτήσεις για την ρευστότητα, για την αντιμετώπιση των κινδύνων και με καλύτερη διακυβέρνηση βλέπουμε ότι η κρίση κατέδειξε τις ανεπάρκειες του συστήματος τα προηγούμενα χρόνια. Επίση, αναλαμβάνουμε δεσμεύσει που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο G20. Οι υπουργοί, οι οποίοι συνεδριάζουν αυτή τη βδομάδα στην Ουάσιγκτον, κ. Κρέιτον, αναφέρθηκε στο ρόλο των προηγούμενων ε, προεδριών, κυρβιακή, πολωνική, δανική, αλλά και την ε, και αυτήν της ε, Ιρλανδίας, ε, που θα ευχαριστήσω. Εδώ επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω προσωπικά τον εισηγητή, τον Ότμαρ Κάρας, ε, που ήταν πρόθυμο και φυσικά ικανό, παράλληλα και του άλλου εισηγητέ, την κυρία Μπόους, τον κύριο Μπούλμαν, Λάμπερτ, Φόρντ, που βοήθησαν τον κύριο Κάρας συμμετείχα σε πολλούς από τους τριμερείς διαλόγους του τελευταίες εβδομάδες και είμαι σε θέση να σας πω ότι πραγματικά πρόκειται για έναν πολύ δυναμικό συμβασμό ο οποίος κατέστη δυνατός λόγω της κατανόησης που επέδειξαν πολλοί εξημών στην εξέβρεση λύσεων. Θα ήθελα να τονίσω κάποια σημαντικά σημεία επί των οποίων το Κοινοβούλιο Πρώτη είναι μια περαιτέρω πρόοδο σε σχέση με την αρχική πρόταση. Ένα θέμα πολύ σημαντικό στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε, ε, μια ιδιαίτερη αναφορά και θα ήθελα να πω ότι και εγώ προειδοποίησα τις ε, ε, Ευρωπαϊκές Αρχές, ναι, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και διάλογο του κ. Ταγιάννη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν οφείλει στο Ευρωκοινοβούλιο την δυνατότητα διαμεσολάβησης ε, της ε, Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Αρχής και την ενίσχυση του ρόλου του Κοινοβουλίου στην διαδικασία έγκρισης τεχνικών κανόνων και ρυθμίσεων υποχρέωση των τραπεζών να υποβάλουν στους επόπτες, στους ουθέους αρχές, τις μη ρυθμιζόμενες ε, απαιτήσει. Αυτό εμπίπτει τη εργασίε που θα υποβάλω στο εντό σύντομου χρονικού διαστήματο. Επίση και μια άλλη σημαντική πρόοδο χάρη στο Κοινοβούλιο είναι αυτό τη διακυβέρνηση τη διαφάνεια των αμοιβών. Ε, η εργασία που έγινε για το Capital Requirement 3 και βλέπω την κυρία Μακάρτη ε, εδώ μέσα στην αίθουσα η οποία συνέβαλε πολύ στην διαφάνεια που προτάθηκε, ιδιαίτερα η πλησίωση των ε, αμοιβών. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται μια στιγμή όπου οι τράπεζες ε, φυσικά αποτελούν τμήμα της κοινωνίας. Δεν βρίσκονται εκτός αυτής, όπως μερικές φορές έχουμε την εντύπωση και μιλάμε για μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Σχετικά λοιπόν με αυτές τις καινοτομίες νομίζουμε ότι έχουμε τα στοιχεία για να προχωρήσουμε σε μια διεθνή συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι η, μοναδική, μόνο ότι είναι η πρώτη που προτείνει κάτι τέτοιο. Πρόκειται λοιπόν για ένα συμβασμό ικανοποιητικό. Όλοι καταβάλαμε προσπάθειε συμπεριλαμβανομένε και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου πιστεύω ότι ο μηχανισμό ε, εθνική ευελιξία δεν έχει ακόμα ε, συσταθεί οριστικά ε, διάλογος με τον εισηγητή αλλά και με εσάς κυρία Μπόλς ε, παραμένει ένα θέμα σημαντικό σχετικά με την δυνατότητα αντιστάθμισης των διαφόρων στοιχείων των ε, συμβάσεων ΛΥΠΟ η Επιτροπή της Βασιλείας θα πρέπει στο μέλλον να προτείνει μια διαβούλευση προκειμένου να εγκρίνει την τελική της θέση στα τέλη του 2013 πιστεύω ότι θα ήταν λογικό και προτιμότερο να μην ε, ε συζητήσουμε τώρα για αυτά τα συμπεράσματα, να τα αφήσουμε για αργότερα, διότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το κείμενο και να αφαιρεθεί μια φράση από το άρθρο 416 γνώμη, που θα ε, απέτρεπε την ε, αντιστάθμιση. Νομίζω λοιπόν κυρίες και κύριοι βουλευτές ότι έχουμε ένα κείμενο ιδιαίτερα σημαντικό ε, αυτό που ονόμασα το single rule book στον τραπεζικό κλάδο και αν εδώ προσθέσετε στο κείμενο ενώ όταν θα είναι λειτουργικό χάρη σε εσάς στις αρχές του 2014 στην εποπτεία των τραπεζών σε επίπεδο ενίας αγοράς ε, χάρη στις νέες αρχές που ιδρύσαμε αλλά χάρη και στην Κεντρική Τράπεζα που από τον ε, Άνοιξη του 2014 θα έχει μια άμεση εξουσία αμεσότερη εξουσία. Στο κείμενο λοιπόν το οποίο θα πρέπει τώρα να ολοκληρωθεί το είπαμε στο Δουβλίνο με τους υπουργού και το, θα θέλω να το επενθυμίσω ή δυνατόν να εγκριθεί κατά τη διάρκεια της Ιρλανδική Προεδρία Το θέμα αυτό, το κείμενο αυτό συζητείται εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Έχουμε στοιχεία τα οποία αν είχαν ε, συσταθεί και τεθεί σε λειτουργία θα είχαν περιορίσει ή παρεμποδίσει την τραπεζική κρίση και δεν έχω κατά νου μόνο την Κύπρο αλλά και άλλες χώρες και οι φορολογούμενοι είναι αυτοί οι οποίοι πέστησαν εδώ και 5-6 χρόνια τις επιπτώσεις λοιπόν ας πάμε στο τέλος ε, για να σε στο σύνολο το αυτό το single ε, rule book χρειάζεται λοιπόν ένα βολονταρισμό για να το πετύχουμε και πιστεύω ότι παράλληλα η ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παίξουν τον ρόλο τους, τον εποπτικό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας ευχαριστώ για τη δέσμευσή σας επί αυτού του σημαντικού κειμένου το οποίο ε, ελπίζω να μπορέσετε να εγκρίνετε σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπαρνιέ. Τώρα έχουμε τους ομιλητές εκ μέρους των ομάδων. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ έχει το λόγο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να λάβουμε υπόψη την σταθερότητα και να την εγγύσουμε τη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ότμα Κάρας για την εξαιρετική αυτή εργασία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για να φτάσουμε σε μια συμφωνία μαζί με άλλους συναδέλφους βεβαίως. Μιλάμε για μεγάλες ε, ε, πρωτοβουλίες και προτεραιότητες του ΕΛΚ. Μιλάμε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές κρίσεις. Και εδώ μιλούμε για τις συστημικές, συστημικές τράπεζες, οι οποίες δεν θα πρέπει να διασωθούν από τους φορολογούμενους. Είναι ύψη της σημασίας λοιπόν, έτσι ώστε οι τράπεζες να μην αναλαμβάνουν υπέρμετρους κινδύνους θα πρέπει οι τράπεζες επίσης να χορηγούν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως ως προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις το θέμα αφορά τις ΜΜΕ και μία νέα βάση για την τραπεζική μας ένωση. Κύριε Επίτροπε, συμφωνώ ότι θα πρέπει να δώσουμε απτή μορφή σε αυτή την τραπεζική ένωση και θα πρέπει η ΕΚΤ να εποπτεύει το τραπεζικό σύστημα. Η συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών της Ιρλανδίας πώς θα πρέπει να ερμηνευθεί ε, ως καθυστερημένη παρέμβαση ή ως έγκαιρη. Επίσης, ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε στην, για την φάση εφαρμογής. Αυτό αφορά και τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων. Θα πρέπει να υπάρξει κάτι συγκεκριμένο και για τον Οργανισμό Εξυγίανσης των Τραπεζών. Σας ευχαριστώ κύριε Βορτμαν Κόλ και τώρα ο κύριος Γκούλμαν για 3,5 λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω και εγώ, και το λέω εκ μέρους της ολυδημοκρατικής μας ομάδας, ότι επετεύχθη πολύ σημαντικό έργο αυτό το κείμενο, ορατό έργο, μάλλον πρόκειται για, το πιο, ε, για την πιο αποφασιστική στράτευση μετά την κρίση για τη μεταρρύθμιση των τραπεζών. Και θα ήθελα προκαταβολικά να κάνω μία παρατήρηση ότι δεν ήταν καθόλου εύκολα το έργο αυτό. Διδαχθήκαμε μάλιστα ότι ε, διαπιστώσαμε μάλιστα ότι τα διδάγματα της κρίσης κάποιοι δεν τα αντιλαμβάνονταν και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορεί να θεωρούν από τις τράπεζες ότι πλήττονται υπερβολικά από αυτές τις διατάξεις. Όχι, φαίνεται ότι στους μεγάλους, στα μέγαρα τα τραπεζικά δεν έχουν αντιληφθεί ποια είναι τα διδάγματα της κρίσης. Και αυτό πολλές φορές θα πρέπει να το πούμε και στα Υπουργεία των Οικονομικών, γιατί θα είχαμε προχωρήσει πολύ, πολύ νωρίτερα αν είχαν συνεργαστεί. Και στα εθνικά λοιπόν Υπουργεία των Οικονομικών βλέπουμε να παραμένει ακόμη ζωντανό το πνεύμα του πρόπερση ουσιαστικά. Γιατί λένε ναι θέλουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα αλλά με την οτροπία του παρελθόντος. Δεν γίνεται λοιπόν. Και γι' αυτό θα ήθελα κυρίε και κύριοι να απευθύνω θερμές ευχαριστίες του Ρότμαν Κάρα τη οφείλω, γιατί ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων και προ ολόκληρη βέβαια την ομάδα των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί δεν ε, συνεργάστηκαν μόνο οι βουλευτέ, αλλά και οι εξαίρετοι ε, συνεργάτες, τα μέλη του προσωπικού που είχαμε στην ε, ομάδα μας και θα ήθελα κύριε Μπαρνιέ να πω ότι προχωρούν όλα αυτά στην νομοθεσία διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν κάμπτεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να δώσει τις ορθές αποφάσεις όχι μόνο εδώ στην ΟΚΑ 4 αλλά και στο θέμα των τραπεζών και στα ε, hedge funds και στις, ε, στο θέμα των οργανισμών αξιολόγησης ε, πιστοληπτικής, ικανότητα, ικανότητας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να ανατρέψει τα πάντα και να εισαγάγει τη σωστή, την ορθή, την απαραίτητη νομοθεσία σε όλους αυτούς τους τομείς, όπως άλλωστε πράττει και εδώ. Και όντως θα χρειαστεί να ε, διατυπώσουμε πολύ πιο αυστηρούς κανόνες για να λειτουργεί το σύστημα σωστά. Χωρίς διαφοροποίηση όμως. Γιατί το, στον δρόμο αυτόν λέμε αυτό ακριβώς ότι όποιος γεννά κίνδυνο θα πρέπει να περιμένει και πιο αυστηρή αντιμετώπιση για να μην επιβαρύνει όλους εκείνους που έχουν μπορέσει να ε, να επιβιώσουμε μέσα στην κρίση που έχουν κάνει καλή δουλειά τις μικρομεσαίες εκείνες επιχειρήσεις που αγωνίζονται και ε, εργάζονται. Άρα λοιπόν θα κάνουμε διαφοροποίηση ανάλογα και με το προφίλ της διακινδύνευσης αλλά και με τα σημεία μόχλευσης, όλα αυτά θα τα δείτε στα κείμενα. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε όμως επιπλέον ε, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις δεν θέλουμε να ε, υπονομεύσουμε τις δυνατότητες για ανάπτυξη νέων και σύγχρονων υποδομών. Αυτά όλα τα έχουμε συζητήσει όπως έχουμε συζητήσει και τις εθνικές ιδιαιτερότητες που απαιτούν απαντήσεις διαφορετικές κατά περίπτωση. Σε αυτό απαντούμε ναι στο βαθμό που δεν, παρα, δεν διαταράσσεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στο βαθμό όπου δεν κινδυνεύει η αξία της δικαιοσύνης και της κατανομής των βαρών. Όπου δηλαδή υπάρχουν πολλές, πολλά κέρδη, εκεί θα υπάρχουν και πολύ πιο αυστηροί έλεγχοι. Η κυρία Μπόλζ έχει το λόγο. Ήταν τεχνική η φύση όλη η διαπραγμάτευση, αλλά το τελικό πακέτο ήταν πολύ καλό. Θα θα ήθελα λιγότερη ρύθμιση και ενίσχυση αντιμετώπισης των παραγόγων προϊόντων. Τα μπόνους βρίσκονται στο προσκήνιο έναντι της άλλης εργασίας και θα πρέπει να υπάρχει ε, εξισορρόπηση της, ε, της αναλογίας παροχής μπόνους, ε, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για παρακινδυνευμένη συμπεριφορά. Ως προς το χρηματοπιστωτικό τομέα βλέπουμε ότι η Ευρώπη έχει πρωταρχικό ρόλο και προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους των ε, βραχυπρόθεσμων δανείων. Επίσης προσπαθούμε να μην ε, εντάσσονται τα hedge funds σε, να, να αντιμετωπίζονται μέσα στα πλαίσια του CVA και έχει μεγάλη σημασία να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες γιατί πολλές φορές ε, δεν υπάρχει ε, δυνατότητα αντιμετώπισης των hedge funds. Και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχουν αποκαλύψεις σε σχέση με το ποιος ακολού, δεν ακολούθησε σωστή συμπεριφορά στην αντιμετώπιση στοιχείων ενεργητικού. Θα πρέπει να βλέπουμε το παρελθόν των τραπεζικών αρχών και των τραπεζιτών. Να δούμε ποια ήταν η συμπεριφορά των παρελθόντο, του παρελθόντος όλων. Και αυτό ε, άρχισε από εδώ θα πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση ως προς, τον, προς αναστολής ε, του, των ε, κεφαλαιακών αρχών και να δούμε πώς ε, θα ενισχύσουμε την εξυγίανση. Υπάρχουν υπολοιπόμενα θέματα, αλλά ως προς την αντιμετώπιση των στοιχείων... Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπόλς. Λάμπερτς παρακαλώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί στην Ευρώπη για να πούν ότι η Ευρώπη δεν κάνει τίποτα για τα δημοσιονομικά. Τουλάχιστον ο κ. Μπαρνιέ δεν πρόκειται να το πει. Ε, είναι ένα μια ε, θέμα πολύ σημαντικό. Ε, αφορά ένα σύστημα πολύ σημαντικό αυτό των τραπεζών, το συστημικό τραπεζ, σύστημα. Λοιπόν, το τραπεζικό σύστημα είναι πολύ μεγάλο για να το αφήσουμε να χρεοκοπήσει και σήμερα πραγματικά επιτυχαίνουμε κάποια κάποιους πόντους, κάποια συν Μιλήσαμε για τις ανάγκες ε, κεφαλαϊκής επάρκειας ε, και τη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτού και της συστημικού κινδύνου. Οι κανόνες λοιπόν που προτείνουμε είναι ζήματα έκτακτης σημασίας ε, και αφορούν να τη διαφάνεια αλλά και τις αποδοχές. Πολλές φορές άκουσα να λέγεται ότι οι αμοιβές δεν είναι το πρόβλημα ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι βρίσκονται στο επίκεντρο και είναι ο πρώτιστος ε, στόχος ε, των συνεπειών που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε λοιπόν τον κανονισμό σε 3 που κάνει το συσχετισμό μεταξύ των σταθερών αμοιβών και των ε, συνδεδεμένων με τις επιδόσεις αποδοχών πιο λοιπόν επαναστατικό είναι το, η έκθεση αναχώρα, το αναφέραμε επανειλημμένα στη συζήτηση. Όχι, η αδιαφάνεια δεν θα πρέπει να είναι ο κανόνα εξάλλου ένας Μια ανταγωνιστική οικονομία απαιτεί τη διαφάνεια και την ισότιμη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων. Αυτό είχα πει και στο παρελθόν και αισθανόμουν όσο τελευταίο φιλελεύθερος ε, ε, πρότεινα τον αθέμητο ανταγωνισμό. Λοιπόν, πώς γίνεται λοιπόν να μπορέσαμε να ε, ε, ε, έχουμε ικανοποίηση πάνω στα δύο σημεία τα οποία θεωρούμε απαραίτητα διότι μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε την αντίσταση των τραπεζών που στήριζαν πολλοί υπουργοί οικονομικών που έπαιξαν το ρόλο του συνηγόρου των τραπεζών μέσα σε μια προσπάθεια που, μάλλον σε μια βούληση που ξέφρασε το κοινοβούλιο μας Ομοφόνο και την, μια κοινή γνώμη η οποία φυσικά ήταν κατά της αδιαφάνεια και των υπερβολικών αμοιβών. Ένα από αυτά τα δύο σημεία ε, εκλείψει, τότε δεν πετυχαίνουμε το στόχο μας Και έτσι οι κανόνε δεν πάνε αρκετά μακριά. Ήδη οι πόροι λοιπόν θα παραμείνουν και αύριο με βάση τα σταθμισμένα ενεργητικό που υπολογίζεται από τις τράπεζε για να ελεξιτοποιήσουν τις απαιτήσει σε κεφάλαια. Γνωρίζω πως από πλευρά ε, Κομισιόν ε, υπάρχουν κάποιες σκέψεις, αλλά δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί. Και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποιους υπουργού οικονομικών που έπαιξαν το ρόλο της αντίδρασης. Θα πω ιδιαίτερα στον Πιέρ Μοσκοβίση ότι το συμφέρον της Γαλλίας ε, δεν συγχαίρεται με αυτό της Μπεν Πέι, της Bank Agricole. Να πούμε στον κύριο Σόιμπλερ ότι τα συμφέροντα της Γερμανίας δεν ε, δεν ε, υπερισχύουν του κοινού συμφέροντος ε, το οποίο και θα πρέπει να υπερισχύσει. Θα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τρεις πρωταγωνιστές αυτού του θέματος. Πρώτα απ' όλα, τη Βρετανική κυβέρνηση μπορεί να φαίνεται παράδοξο μετά από την τσακωμό που είχαμε για τα αμοιβές, αλλά σήμερα ο κίνδυνος ε, τον οποίο δημιουργούν οι συστημικές τράπεζες στην οικονομία μας και στις κοινωνίες μας ε, είναι κάτι το οποίο ε, με το οποίο συμφωνεί και η Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστώ προσωπικά τον Μισελ Μπαρνιέ που είναι ο κινητήρας, κινητήρας δύναμη από πλευράς Κομισιόν για την ε, διευθέτηση των, των προβλημάτων του ιστορικού κλάδου. Ε, ε, έχουμε έναν, έχουμε έναν επίτροπο ο οποίος υποστηρίζει την εποπτεία και είναι κάτι το πολύ θετικό να έχουμε σένα ως αρμόδιο επίτροπο και ευχαριστώ επίσης και τον Νότ Κάρας που μπόρεσε να ξεπεράσει τις κομματικές διαφορές και να υποστηρίξει το γενικό συμφέρον και ειδικά το συμφέρον και την ε, θέση του Κοινοβουλίου. Διότι όπως λέμε ένας, πολιτικό πολιτικός πρέπει να γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι του. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φόρντ έχει το λόγο. Ε, ο τραπεζικό τομέα έχει όλο και πιο διεθνή χαρακτήρα, πιο παγκόσμιο χαρακτήρα και γι' αυτό χρειάζεται αντιμετώπιση και σε παγκόσμιο επίπεδο για να υπάρχουν ισότιμε συνθήκε ανταγωνισμού. Έγιναν λοιπόν πολλέ προσπάθειε για την προσαρμογή στι παγκόσμιε διατάξει και προδιαγραφέ των ευρωπαϊκών ε, προδιαγραφών, ωστόσο δεν ολοκληρώθηκαν αυτές οι προσπάθειες και έτσι δεν είναι ευθυγραμμισμένο το δικό μας πακέτο με τις προδιαγραφές της Βαρκελόνης. Εμείς θέλουμε ως ομάδα να προστατεύονται και τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου, ε, να μην ε, ζημιώνεται δηλαδή από την ε, καταβολή των αμοιβών στους τραπεζίτες εις βάρος της καταβολής μερισμάτων ή επιστροφής των χρεωστουμένων. Και γι' αυτό είδαμε και τα δεινά που αντιμετώπισε η Κύπρος πολύ πρόσφατα, επειδή δεν, δεν ίσχυαν αυτές οι διατάξεις. Η... Δε ε, συνθήκες για την ασφάλιση των τραπεζών ε, δεν ακολουθούν τις παγκόσμιες προδιαγραφές Χρειάζεται λοιπόν να προχωρήσουμε, να εργαστούμε ακόμη περισσότερο όλοι εδώ στο Κοινοβούλιο, ώστε να εξασφαλίσουμε εγγύησεις και για, τους, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για, τις, ε, για τη διακυβέρνηση, την εταιρική, ε, για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και της ε, ορθής λειτουργίας τους. Έχουμε προσπαθήσει πολύ να πείσουμε ότι οι υψηλέ προδιαγραφές έχουν μεγάλη αξία και θέλουμε να πείσουμε και τι κυβερνήσει. Δεν πρέπει λοιπόν να χαθούν αυτές οι προσπάθειε. Ω προς τις αμοιβέ ε, των τραπεζιτικών Ξέρουμε ότι χρειάζεται παγκόσμι, σε παγκόσμιο επίπεδο αυτών και εμεί έχουμε κάνει προτάσεις ώστε να είναι πιο μακροπρόθεσμη η θεώρηση αυτών των αμοιβών αλλά να μην γίνεται προκαταβολικά η καταβολή του, των πρίμα. Εμείς δεν θα κατα... Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Μπλουμ. Νομίζω ότι εδώ προσπαθούμε να πούμε ότι ελπίζουμε θριαμβεύει η ελπίδα έναντι της Πύρας. Το πρόβλημα που έχουμε είναι ένα λανθασμένο τραπεζικό σύστημα, ένα κατακαιρματισμένο σύστημα όπου οι τραπεζίτες δανείζουν χρήματα που δεν έχουν. Στις ΙΠΑ το 1850 αυτό επέσυρε θανατική ποινή και το να μην υπάρχει ρύθμιση είναι ένα είδος ρύθμισης και έτσι φτάσαμε σε μία άλλη καταστροφή και τίποτα δεν θα μας σώσει από μία επικείμενη καταστροφή και δεν ε, θα έχουμε παρά καταστροφές διότι θα πρέπει να υπάρχουν τράπεζες ε, σε σχέση με την παροχή ε, ρευστότητας και παροχής αγαθών. Θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κλειδονισμούς. Τι θέλουν οι άνθρωποι, οι άνθρωποι θέλουν τα χρήματά τους πίσω και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κατάλληλα. Μιλάμε για τα μπόνους των τραπεζών. Εδώ έχουμε, έχουμε εγκληματική δραστηριότητα των ε, τραπεζιτών και κανένας δεν ε, έχει σταλεί στη φυλακή. Δηλαδή πολλά ε, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια στερλινών έχουν φύγει από τις τσέπες των φορολογούμενων και κανένας δεν έχει πληρώσει. Θα πρέπει να μην έχουμε λοιπόν τόσο μεγάλη ρύθμιση. Μιλάμε για ε, τύπωση χρημάτων. Θα ήθελα μερικούς κεντρικούς ε, τραπεζίτες ε, στη φυλάκιση, γιατί όταν τυπώνουμε χρήματα, τι κάνουμε, παραχαράσουμε. Είναι παράνομο. Ας δούμε λοιπόν προς τα έσω. Να δούμε δηλαδή τι κάνουν οι κεντρικοί τραπεζίτες, οι πολιτικοί και οι οποίοι δρούν κατά των φορολογουμένων. Ας τους δούμε στις ε, φυλακές λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος δύο μισή λεπτά. Υπάρχει μια μπλε κάρτα. Ο πρόεδρος, δυστυχώς δεν έχουμε χρονικό περιθώριο για μπλε κάρτες. Ο κύριος κλούτε. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Τις τελευταίες ημέρες ε, μίλησαν κάποιοι συνάδελφοι για επανάσταση με την εισαγωγή αυτή τη προτάσεω ο 4. Εγώ δεν θα έφτανα μέχρι εκεί, αλλά θεωρώ ότι πραγματοποιείται ένα πολύ σημαντικό βήμα. Ανασυγκρότηση και σταθεροποίηση του τραπεζικού χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το αποτελεσμά τη και θα πρέπει να συγχαρούμε τον κύριο Τμαρκάρα, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά επί τη βάση των προτάσεων του Επιτρόπου κυρίου Μπαρνιέ. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε από πλευρά μα. Ιδιαίτερω υποστηρίζουμε την ε, εξασφάλιση ενός ε, ε, διαφοροποιημένου τραπεζικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις ε, τράπεζες αποταμίευσης, τα ταμιευτήρια σε περιφερειακό επίπεδο δεν μπορούμε να τις εντάξουμε μέσα στην έννοια των μεγάλων ε, τραπεζών. Οι συνεταιριστικές τράπεζες ή ταμιευτήρια έχουν επιδείξει μεγάλη σταθερότητα στις ε, περιόδους της κρίσεως, έχουν σταθεί σταθερή αρρωγή στον μικρό και μεσαίο επιχειρηματία και θα πρέπει ασφαλώς να τις διαφοροποιήσουμε από τους άλλους ε, τραπεζικούς οργανισμούς. Ο κύριος Μπούλμαν ήδη επεσήμανε κάποια στοιχεία. Επίσης, η ρύθμιση για τα μπόνους και τα πριμ είναι για μένα αποδεκτή και τη δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν δέχθηκε την αρχική πρόταση στο Συμβούλιο. Μια ρύθμιση ένα προς ένα η οποία θα ήταν πολύ πιο καλή και πιστεύω πολύ πιο αποδεκτή για τον πολίτη και ψηφοφόρο. Ένα σημαντικό θέμα πάντως πραγματοποιήθηκε παρόλα αυτά. Επίσης, την ε, προσφορά ιδίου κεφαλαίου. Εμείς είχαμε στήσει 18% στη δική μας πρόταση. Άλλοι είπαν ότι δεν είναι δυνατόν αυτό. Άλλοι ζήτησαν ε, να είναι 15% το ποσό αυτό, το οποίο δεν απήχε τόσο πολύ από τη δική μας αρχική προσφορά και ως εκ τούτου μπορούμε να τη δεχθούμε. Κάποιες άλλες επικριτικές ε, ε, παρατηρήσεις για το ποσοστό ε, μόχλευσης, leverage ratio, ε, στο οποίο θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να εισαχθεί η αρχή των κατεξουσιοδότηση πράξεων. αλλά θα έπρεπε να παραμείνει στην συναπόφαση η ρύθμιση αυτή. Εμεί θέλαμε πάνω απ' όλα να υποστηρίξουμε τις μικρές τράπεζες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κλούτε. Ο κύριος Σέλστρα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι κεντρικέ τράπεζες ε, θα έπρεπε να ε, ελέγχουν ιδιαίτερα τους ροές μεταξύ τραπεζών, διότι η, η δημιουργία χρήματος ε, δημιουργεί πληθωρισμό. Ξέρουμε ότι κάποιες τράπεζες μπορούν να ανταγωνιστούν, άλλες όχι. Αυτός είναι ο οικονομικός δαρβινισμός. Η οικονομική ζωή από ό,τι ξέρουμε εξαρτάται από τις ε, τράπεζες αλλά με τη νέα αυτή οδηγία οι τράπεζες χάνουν κάποιες ε, ε, κάποια προνόμια και όταν μια τράπεζα δεν πάει καλά τότε το προσωπικό απολύεται και η τράπεζα χρεοκοπεί, κλείνει. Εμείς εδώ δεν κάνουμε διαφορά ανάμεσα στις ε, χώρες. Λέω ε, ένα παράδειγμα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αντικαταστήσει κάτι το εθνικό με ε, μια διαδικασία υπερεθνική. Αυτό νομίζω ότι είναι καλό. Μία τράπεζα λοιπόν η οποία την χάνει σωστή διαχείριση, δεν λαμβάνει υπέρμετρους κινδύνους. Αυτές οι ευρωπαϊκές αποφάσεις νομίζω ότι θα προλάβει Παρόμοιε καταστάσει. Μια καλύτερη διαχείριση των πιστώσεων θα μας ε, οδηγήσει στην αποφυγή της κρίσης. Αλλά έχω την εντύπωση πω ε, εδώ προθούμε να ε, ρυθμίσουμε τα πράγματα ενώ τα, η κατάσταση έχει, έχει καταστεί πραγματικά τραγική. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σέλστρα και δεν μπορώ δυστυχώς να δεχθώ μπλε κάρτα, ειδικά σε εκείνους που έχουν ήδη ε, μιλήσει ή που είναι ήδη γεγραμμένοι στον κατάλογο. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Μπάλτς να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ότμαν Κάρας, τον εισηγητή του Κοινοβουλίου και να τον συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά του αλλά βέβαια και τους και οδησηγητές που έχουμε συμπράξει αυτήν. Με την έκθεση αυτή το Κοινοβούλιο μιλάει με πολύ πιο αυστηρούς κανόνες για τη ρύθμιση της, ε, του τομέα των αγορών, των τραπεζών, συγγνώμη, προς το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Πιστεύω ότι αυτοί οι ουσιώδεις για τη συζήτηση κανόνες και τα μπόνους, τα πριμ των ε, ε, στελεχών θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποφασιστικά. Ε, η κρίση μας έχει δείξει ότι πρέπει να αναλαμβάνουμε αποφασιστικά βήματα και στην προκείμενη περίπτωση το επιτυγχάνουμε με μια δίκαιη αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν κοιτάμε μάλιστα ποια είναι η νομική μορφή, αλλά τι είδους κεφάλαια διαχειρίζεται ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και δι' των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο παράγων κινδύνου για τις μικρές και μεσαίες πιστώσεις πέφτει στα 50% και ως εκ τούτου μειώνεται αντίστοιχα και η, προσφορά, η απέτηση για προσφορά ιδίων κεφαλαίων. Η έκθεση αποτελεί μεγάλη επιτυχία για ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπάλτς. Η κυρία Μακάρτη, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Κάρα και την διαπραγματευτική του ομάδα. Το 2010 είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε για τη θέσπιση κανόνων ε, σχετικών με τα μπόνους των στελεχών που θα μπορούσαν είτε να μην καταβάλλονται ε, να καθυστερεί η καταβολή τους, να ανακτώνται και να αμφισβητούνται. Τώρα βλέπουμε ότι έχουμε προχωρήσει σε ένα ανώτατο επίπεδο 1 προς 1 ή 1 προς 2 για τα μπόνους και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε έτσι να θέσουμε ένα τέρμα σε ένα αφόρητο σύστημα τραπεζικό όπου έχουμε τράπεζες με 2,5 εκατομμύρια ε, απώλειες, 1,5 εκατομμύριο σε πρόστιμα και ακόμη 1,5 εκατομμύριο σε επιβαρύνσεις Λίμπορ και όμως παρόλα αυτά μπορούν να ε, καταβάλουν πολύ σημαντικές ε, ε, πολύ σημαντικά μπόνους στα στελέχη του, στα νότατα στελέχη του. Είναι μεγάλο όνειδος αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις τράπεζες του τραπεζικού του πολιτική. Αυτό όμως ε, ο πολίτης το καταδικάζει. 76% ήταν οι πολίτες οι οποίοι το 2010 θέλανε πιο αυστηρή νομοθεσία και ανώτατα επίπεδα στα μπόνους. Και ενώ μπορεί να κερδίζει ένας χρηματιστής ε, 5.000 λίρες ε, το μήνα μπορεί ε, το πριν που παίρνει ακόμα να φτάνει και τις 80.000 τις 8.000 επιπλέον το μήνα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να δεχθεί ο πολίτης και πρέπει πλέον να θέσουμε ένα τέρμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος, η κυρία Γκουλάχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας την Επιτροπή και το Συμβούλιο και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο διότι ο Ότμαρ Κάρας και η ομάδα του δείξανε ότι όταν εργαζόμαστε τόσο και τόσο καλά μπορούμε να φτάσουμε σε απτά αποτελέσματα. Το λέω γιατί δεν συμμετείχα ε, σε αυτή την ομάδα, άρα δεν υπάρχει ίδιο συμφέρον. Θα ήθελα να τονίσω δύο σημεία ως προς την προστιθέμενη αξία του Κοινοβουλίου. Πρόκειται για την πιστοληπτική μας ικανότητα και τη χορήγηση δανείων προς τις ΜΜΕ. Δεν μιλάμε λοιπόν παρά για επενδύσεις και ανάπτυξη, καθώς και διαφάνεια, που είναι κάτι το οποίο ε, δεν είναι ανώδυνο σε αυτό το κείμενο, αλλά μπορεί να αλλάξει πολλά όχι μόνο για τις ε, επιχειρήσεις, αλλά εκεί που υπήρχε αδιαφάνεια και μπορούσαν να γίνουν ύποπτες πράξεις. Ε, ελπίζω να τα καταφέρετε, κύριε Επίτροπε. Ε, κρατήστε γερά. Αυτό που έχει σημασία είναι η εξυγίανση και να θέσετε το Συμβούλιο ενώπιον των ευθυνών του. Υπάρχουν υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν να ακολουθήσουν το Συμβούλιο στις αποφάσεις του παρελθόντος Ιουνίου, δηλαδή μια πραγματική τραπεζική ένωση. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κουλάρ. Στρέτσεκ, ένα λεπτό. Ε, Κυρίες και κύριοι, η σημερινή συζήτηση αφορά ε, δύο διαφορετικά θέματα, τις υψηλές προσδοκίες από τη μία πλευρά και τις ανησυχίες που εκφράζονται. Δεν ε, υπόθηκαν πολλά ως προς τις ανησυχίες. Οι υψηλές προσδοκίες σημαίνουν ότι αν είχαμε περισσότερη ρύθμιση δεν θα είχαμε κρίση ούτε οικονομικούς κλειδονισμούς. Δεν το συμμερίζομαι αυτό, αλλά καταλαβαίνω ότι κατέχει δεσπόζουσα θέση στο σώμα. Από την άλλη πλευρά όμως, η υπουργό Κρέιτον μας ε, έπεισε ιδιαίτερα, ήταν ιδιαίτερα πιστική όταν είπε ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι δεν ρυθμίσαμε κατά τρόπο ώστε η οικονομία να διαθέτει τους πόρους που έπρεπε. Δεν τους διέθετε. Επίσης, δεν θα πρέπει να υπάρξει ρήξη με τους εθνικούς ρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ. Μοργάν, την άμιση λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σίγουρα οι τράπεζες είχαν μια τεράστια ευθύνη για την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Κάθε μέτρο το οποίο θα μας βοηθήσει στο να μην επανελειφθούν παρόμοιες καταστάσεις θα πρέπει να στηριχθεί. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από ισχυρέ τράπεζες ε, και από πολίτε υπεύθυνου. Δεν είναι δυνατόν οι φορολογούμενοι να είναι αυτοί οι οποίοι να προστρέχουν σε βοήθεια ε, των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ε, πιο απλή λύση για μένα θα ήταν μια πρόταση που επαναλαμβάνω εδώ και χρόνια. Μια σαφή ένα σαφή διαχωρισμό ανάμεσα σε εμπορικέ τράπεζε και τι τράπεζε τι επιχειρηματικέ. Ε, ένα νόμο του Αμερικάνικου από το 1932 λειτουργήσε με τα τέλη του δεκαετία του 1990 και δεν νομίζω ότι ήταν απλή σύμπτωση που από την κατάρρισή του πολλαπλασιάστηκαν οι, τα προβλήματα στον τραπεζικό τομέα και οι χρεοκοπίες. θα έπρεπε να θέσουμε λοιπόν ένα τέλος στις αμοιβέ και στα μπόνους των managers είναι λοιπόν απαράδεκτο η, η, η δημιουργία αυτής της κρίσης να ε, αμείβονται. Πριν από ένα χρόνο ο τότε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος έφυγε από την τράπεζα Μότερντε Πάσκη με ένα μπόνους 5 εκατομμυρίων και τώρα βλέπουμε την καταστροφή που δημιούργησε σε αυτή, με αυτήν την μεγάλη τράπεζα. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι να καταργήσουμε αυτό το σύστημα, κάτι το οποίο ενδεχόμενα να βοηθήσει στο να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μορκάντη. Ο κύριο Σαρκουράκη ένα λεπτό. Η αύξηση τη κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στόχο την εξυγίανση δήθεν του συστήματο ώστε να μην πληρώνει φορολογούμενοι. Οι διπανοκρουσίε για την μείωση δήθεν των πόνου των διευθυντικών στελεχών που όντω είναι πρόβλημα Αποσκοπούσαν να συγκαλύψουν το γεγονό ότι η αιτία τη καπιταλιστική κρίση δεν είναι η ανεύθυνη συμπεριφορά κάποιων τραπεζιτών αλλά η υπερσυσσόρευση κεφαλαίων. η ευρωπαϊκή ένωση κυβερνήσει και μονοπόλια τσακίζουν τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων για να διασώσουν την κερδοφορία των καπιταλιστών καταστρέφουν την εργατική δύναμη με 27 εκατομμύρια ανέργου που αυξάνουν. Για να βγει όμω το καπιταλιστικό σύστημα από την κρίση χρειάζεται να προκληθεί σε μεγάλη έκταση η καταστροφή κεφαλαίων. Αυτό οξύνει του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού, όπω είδαμε στου G20, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα άλλα εμπεριαλιστικά κέντρα. Αυτέ τι συγκρούσει εκφράζουν ο κανονισμό και η οδηγία πρώτα βήματα για τη συγκρότηση του μηχανισμού τη Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Μόνο οι πολύ μεγάλε τράπεζε θα μπορούν να έχουν τη νέα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ενώ οι μικρότερε θα είναι το αντικείμενο εξαγορών και συγχωνεύσεων. Θα έχουμε γιγαντέου σχηματιστικού ομίλου που μεγαλύτερη επιθετικότητα θα εντείνουν την εκμετάλλευση του εργαζόμενου λαού και θα απομυζούν τι καταθέσει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτιν για μισή λεπτό. Σου υποβάλλω τα σέβη μου, Ότσμαρ. Έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά, επιμελή δουλειά και σαν το σκιουράκι έφερες πολλά πολλά φουντουκάκια μέσα στη φωλιά. Αλλά θα πρέπει να πω ότι λείπουν μερικά φουντουκάκια και εγώ από πλευρά μου το διαπιστώνω ως καλός Ευρωπαίος, θα έπρεπε τα μπόνους των τραπεζιτών να περιοριστούν ακόμη περισσότερο, να καλύψουν και την διαχείριση κεφαλαίων και θα έλεγα επίσης ότι θα έπρεπε να είναι πολύ πιο δεσμευτικό το ποσοστό ή ο λόγος της μόχλευσης. Και τι είναι ήδη θετικό το ότι υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του επιχειρησιακού μοντέλου και του κινδύνου. Αλλά γνωρίζεις πολύ καλά ότι μένει το σκληρό καρύδι που πρέπει να σπάσουμε, να ανοίξουμε την, ε, τον διαχωρισμό μεταξύ των επιχειρηματικών, επενδυτικών τραπεζών και των εμπορικών τραπεζών. Και εδώ ακριβώς είναι ο μεγάλος κίνδυνος και η δυσκολία ότι μπορεί να αναπτυχθεί αυτός ο κίνδυνος όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται ο φορολογούμενος εν τέλει από τα λάθη τα επενδυτικά των μεγάλων τραπεζών. Ευχαριστώ πολύ για μισή λεπτό ο κύριος Στόρογιαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Ότμαρ Κάρας και όλους τους σκιώδεις για αυτή την εξέχουσα εργασία ως προς τις δύο εκθέσεις, την προληπτική εποπτεία για τα πιστοτικά ιδρύματα και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Οποιαδήποτε ε, αρχική ε, αποτίμηση ήταν, αποτέλεσε υποτίμηση του κινδύνου. Εγώ θα υπερψηφίσω τις δύο εκθέσεις διότι υπάρχουν όρια για την μόχλευση, υπάρχουν οροφές για τα μπόνους και δημιουργούν τα κατάλληλα κίνητρα για τα πιστοτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων να επιστρέψουν προς την πραγματική οικονομία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να συγχαρώ τον εισηγητή Κάρα ε, και την διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου που κατόρθωσε να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα που είναι οι ελλείψεις του τραπεζικού συστήματος που οδήγησε σε μια πανάκριβη πολιτική δίχως προηγούμενο. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα ε, των ε, πιστώσεων και την, πρόθεση ε, ρυθμίσεων για τα κεφαλαϊκές απαιτήσει των τραπεζών, να ενισχύσουμε την διακυβέρνηση και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα ε, κατάλληλων κινήτρων. Η πρωτοβουλία αυτή ε, αναφέρεται στις δεσμεύσεις που έλαβε το G20 για ένα ισχυρότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα και την αναθεώρηση των κανόνων της Βασιλείας 3. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένας κανονισμός για την ενιαία εφαρμογή των κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μια οδηγία που βελτιώνει την διακυβέρνηση ε, και την εποπτεία. Η συμφωνία έχει τρεις πτυχές πολύ σημαντικές. Αφορά 8.000 τραπεζικά ιδρύματα, με διαφορετική αντιμετώπιση, στηρίζει την πραγματική οικονομία και αναζητά την ορθή εφαρμογή σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω ότι στηρίζει μια αλλαγή νοοτροπίας που όταν θίγει το ζήτημα των σταθερών αμοιβών και των μεταβλητών και αναφέρεται σε λογιστικούς κανόνες αναχώρα και εισαγάγει ε, ε, ευελιξία και την, για την αποφυγή των ε, συστημικών κινδύνων. Η, κανονιστική ρύθμιση θα πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σάντσος Πρασέντο. Κύριο Σμίτη έχει το λόγο. οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερους αναστολής για να μην, και να μην αναλαμβάνουν τόσο μεγάλους κινδύνους. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν οροφές των πόνους διανόμου. Ε, πίστευα ότι αυτό θα επιληθεί από τις τράπεζες καθεαυτές, αλλά φαίνεται ότι κοφεύουν οι τραπεζίτες ως προς αυτό το δημόσιο ε, λόγο. Χαίρομαι διότι το Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρότασή μου να αλλάξει η διαδικασία διορισμού στα διοικητικά συμβούλια. Ε, θα πρέπει σε κάθε τράπεζα να υπάρχει τουλάχιστον μία γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτό θα πρέπει να επιβληθεί. Πρόκειται για μία οδηγία που θα περάσει από την Επιτροπή Οίκων για γυναίκες, για ύπαρξη γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό κύριος Καμάλ. Πρόεδρε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Είναι βέβαια ευπρόσθετο γεγονό ότι καλούμε τι τράπεζε να κάνουν πιο καθαρή, ε, καθαρού συλλογισμού και πιο ε, καθαρές δουλειές. Αλλά αυτό θα μπορούσε να το έχει ρυθμίσει αυτόματα η τράπεζα, το τραπεζικό σύστημα και θα μπορούσαν ε, χωρίς ε, να επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος τράπεζες να έχουν εξηγενθεί. Ε, πρέπει ωστόσο να αναθέσουμε, να να εξασφαλίσουμε ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη οι τράπεζες για τα σφάλματα τους, είτε άμεσα είτε έμεσα και να έχουν τη δυνατότητα να προβλέψουν ε, του κινδύνου ώστε να δημιουργούν αποθεματικό ασφαλεία. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το εξασφαλίσουμε. Η Βασιλεία 1 και 2 προφανώ δεν αρκούσαν ω ρυθμίσει. Φαντάζομαι ότι ούτε και τη τρίτη εκδοχή του θα αποδειχθεί επαρκή. Χρειάζεται να βγούμε από το σύστημα των ε, απλών ε, αποφάσεων θα πρέπει να κάνουμε πολύ πιο ουσιαστική δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάγκεν έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η ΟΚΑ 4, η Βασιλεία 3 είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος τράπεζες και κυρίως όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, αλλά δεν αποτελεί το ε, τελευταίο βήμα, είναι μόνο ένα βήμα στην πορεία αυτή Ευχαριστώ τον κύριο Κάρας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολύ σκληρή δουλειά, άντα τριμερείς διαλόγους ε, σε αυτά τα δύο χρόνια κολυσιεργούσε όχι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αλλά το Συμβούλιο. Στο βαθμό αυτό λοιπόν είναι καλό το γεγονός ότι μπορούμε να έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που επιτυγχάνονται τα σημαντικότερα σημεία, δηλαδή ε, πιο ενισχυμένα κεφάλαια για τις τράπεζες, ευθύνες, περιορισμός των πόνους, Παραμένουν όμως εκρεμή ζητήματα όπως ε, η παγκόσμια, σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμογή αυτών των διατάξεων, εάν συμπράξουν οι μεγάλοι εταίροι όπως οι ΗΠΑ, το ζήτημα του μηδενικού κινδύνου που δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Τρίτον, οι ρυθμίσεις για τα μπόνους θα πρέπει πολύ γρήγορα να ε, υλοποιηθούν και τέταρτον περιμένουμε νέες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμπλήρωση των ρυθμίσεων ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Μπέρες, για μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αγαπητέ συνάδελφε, κύριε Σιγητά, ε, η ρύθμιση για πετήσια ίδια κεφάλαια φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, πρώτο καθεδρία και στην πρώτη γραμμή των αγώνων. Έτσι, η Βασιλεία 3 την πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος μια σειρά από διαπραγματεύσει που κράτησαν πάνω από 20 μήνες μετά την 20η ε, Ιουλίου του 2011 και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και σε όλα τα άλλα ζητήματα τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικού τομέα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν έχει δραματίσει ένα πλήρη ρόλο ω συνομοθέτη, ενώ τα κράτη-μέλη για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προτιμούσαν να υπεραμείνονται θέσεων στρεβλών ως προς τα ίδια κεφάλαια, το καθένα σκεπτόμενο τα δικά του τραπεζικά συστήματα. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα σύστημα απαραίτητο για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία ενός θεναρού τραπεζικού συστήματος που θα στηρίζει την πραγματική οικονομία. Ταυτόχρονα όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμενε και εισήγαγε ε, πολύ πιο δεσμευτικούς κανόνες όσον αφορά τα μπόνους των τραπεζιτικών ώστε να μην είναι τερατώδη πλέον και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τη γαλλική κυβέρνηση η οποία υπερασπίστηκε στο Συμβούλιο τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιμέτωπη με την Βρετανική κυβέρνηση. Όπως άλλωστε εισήγαγε με τις προσπάθειές της και μια σειρά από κανόνες διαφάνειας. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα κύριε Πρόεδρε όταν ολοκληρωθεί αυτό το θέμα και ξεκινήσει η πραγματεύση με τις Ηνωμένες Πολιτείες κύριε Βουαρνιέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αν δεν απαιτήσετε την αμοιβαιότητα στον τομέα αυτό φοβούμαι ότι αυτέ οι ε, συμφωνίες θα είναι ε, ανύπαρκτες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κλίντς για ένα λεπτό. Ε, πάνω στην κρίση ήταν σαφές ότι χρειαζόταν να θεσπιστούν οι βασικές αρχές για ίδια κεφάλαια, ένα μηχανισμό εποπτείας και ένα μηχανισμό διαχείριση κρίσεων. Αυτά τα τρία πράγματα που χρειάζονταν πέρασε πολύ καιρό όμω με τι διαπραγματεύσει και τώρα έχουμε ένα σημαντικό βήμα με τι απαιτήσει για, ε, για τα ίδια κεφάλαια ανεξαρτήτως ε, τη νομική μορφή των τραπεζών που εξασφαλίζει και περισσότερη διαφάνεια και καλύτερε συνθήκε για υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πιστώσει. Αλλά υπάρχουν άλλα θέματα όπω τα κρατικά ομόλογα ε, που αναφέρθηκαν νωρίτερα δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιε ελάχιστε προδιαγραφές τα κρατικά ομόλογα και την έκδοσή τους. Δεύτερον, η δυνατότητα τα κράτη-μέλη να θεσπίζουν ε, ε, ε, τα, τα ύψη των ε, κεφαλαίων μόχλευσης δεν μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ε, στρέβλος των αγορών εντός ευρωπαϊκής αγοράς και στρέβλος του ανταγωνισμού σε επίπεδο τόσο ευρωπαϊκό όσο και διεθνές. Και τελευταίο σημείο, χρειάζεται να αλλάξουν νοοτροπίες της, στον τραπεζικό τομέα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κλίντ, ο κύριος Φέιο τώρα. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να πω επί του θέματος αυτού ότι φτάσαμε σε ένα πολύ καλό κείμενο σε σχέση με τα πιστοτικά ιδρύματα αλλά και γενικότερα σε μία τέτοια δύσκολη χρονική στιγμή οι τράπεζες θα πρέπει να υπηρετούν την οικονομία και τα πρόσωπα, επιτρέποντας επενδύσεις που θα οδηγήσουν στην ανόρθωση της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Τη στιγμή που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι η Ευρωζώνη είναι το επίκεντρο της παρούσης κρίσης, της παρούσας κρίσης θα πρέπει να δώσουμε και την κατάλληλη απάντηση. Δηλαδή να έχουμε πιο ε, στεναρή στάση ως προς τις τράπεζες, οι οποίες να είναι πιο εύρωστες. Η τράπεζα μπορεί να είναι μοχλός ανάπτυξης και φτάσαμε σε ορισμένες κοινέ αρχές για την καλύτερη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Όμως η Τραπεζική Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει. Χρειαζόμαστε κατάλληλους κανόνες για την εξυγίανση των τραπεζών και τις εγγυήσεις των καταθέσεων. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να έχει τον τελευταίο λόγο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νότ Μαρκάρας για την εξαιρετική του εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μισή λεπτό, κύριο Σκαδράουι. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Εξ αρχής ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την ομάδα διαπραγμάτευσης. Αυτό το νομοθετικό πακέτο αποτελεί έναν τρόπο διευθέτησης της κρίσης του τραπεζικού τομέα και αποσόβησης μελλοντικών κρίσεων. Σε σχέση με τις οροφές τα μπόνους, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πιο σωστό ε, μια σωστή αντιμετώπιση για την αντιμετώπιση κινδύνων και ε, οι απαιτήσει ε, κεφαλαιακής ανάπτυξης δείχνουν ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερους αναστολής. Θα έχουμε λοιπόν μεγαλύτερη διαφάνεια και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Τα μέτρα αυτά εξαρτώνται από μία σειρά άλλων ζητημάτων. Η Επιτροπή θα προωθήσει ισχυρή εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο εγγύς μέλλον αναμένουμε προτάσεις για ένα ταμείο εξυγίανσης των τραπεζών έτσι ώστε οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν κινδύνους και δυσκολίες ως προς τον ε, τομέα των ε, τραπεζών θα πρέπει να αποσοφήσουμε οποιαδήποτε μελλοντική κρίση. Ευχαριστώ πολύ. κύριε Τάισερ, λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κρίση ε, δεν έχει περάσει και η εμπιστοσύνη δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα. Αλλά ε, εργαζόμαστε σκληρά, ευτυχώς εξάλλου και πετυχαίνουμε και κάποια πρόοδο. Το βλέπουμε σήμερα με το, ντοσχέ το φάκελο που μας έχει ε, με το οποίο, τον οποίο συζητάμε και έχουμε ενώπιον μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κάρας για τον όλη τη δουλειά μας επέτρεψε να προχωρήσουμε. Αυτό το νομοθετικό πακέτο, αυτή η νομοθετική δέσμη, ε, μας επιτρέπει σήμερα να καθορίσουμε μια σειρά από στοιχεία έτσι ώστε να βοηθήσουμε τον οικονομικό κλάδο και να αποφύγουμε ιδιαίτερα κάποιες ε, βραχυπρόθεσμες συμπεριφορές. Ε, το χρηματοπιστωτικό σύστημα ενισχύει, η οικονομία ε, έχει νέες ευκαιρίες και θα υποφεληθούν οι πολίτες και οι αποταμιευτές οι ε, κανόνες ε, πρέπει να υπάρχουν αλλά χρειάζεται να εφαρμόζονται κιόλας. Ε, απαιτείται εποπτεία. Είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε τις ψωχείς μέρες και εβδομάδες να μπορέσουμε να βασιστούμε σε εσά κύριε Μπαρνιέ προκειμένου να συνεργαστούμε μαζί σας και με την Κεντρική Τράπεζα. Άκουσα τώρα κάτι από την κυρία Φορτμανκόλ και θέτω το θέμα στο Συμβούλιο και την Κομισιόν. Να εφαρμόσουμε τον αφασιστό Δουβλίνο και πώς θα εγγυηθούμε τις καταθέσεις. Ελπίζω να μπορέσουμε να το πετύχουμε μέχρι το τέλος της θητείας. Ευχαριστώ. 1,5 λεπτό κύριε Σπαλώνε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ τον ε, Κάρας και όλους τους σκιώδες ηγητές ε, για αυτήν την εξαιρετική εργασία που έκαναν εξάλλου οι προκλήσεις που είχαμε από την κρίση του 2008 απέτησε μια ε, αναθεώρη, πλήρη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήματος και η οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλόν αυτής της μεταρρύθμισης οι κανόνες της Βασιλείας 3 θα καταστήσουν τις τράπεζες μας πιο ε, ε, ε, πιο αποτελεσματικές και πιο ισχυρές, πιο εύρωστες. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη τον τροπολογία του supporting factor, το οποίο έχει ζωτική σημασία για να αποφύγουμε στρέβλωση των πιστώσεων. Θέλουν, πρέπει να προωθήσουμε την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελέγχουμε κάποιους περιορισμούς στο χρέος και τα κρατικά ελλείμματα. Αλλά αν θα πρέπει να έχουμε ε, ε, καλά δημοσιονομικά στοιχεία θα πρέπει να αποφασίσουν οι κυβερνήσεις να ασχοληθούν με την ανάκαμψη, με την ανάπτυξη. Θα πρέπει να ασχοληθούν με την οικονομική ανάκαμψη υπέρ της ε, και τη στήριξη της ε, πραγματικής οικονομίας. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνουμε και τις πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις, βοηθώντας τις ε, στο να κάνουν περαιτέρω επενδύσεις και να αυξήσουν την εργία δεν απευθύνουμε μάλλον στον κύριο Μπαρνιέ για να κάνει κάτι προσπάθεια για να αυξήσουμε το όριο για να ε, υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άρα της ε, ε, εργασίας για τις αποσχόλησεις. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φέρμπερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι κυρίε και κύριοι, πρέπει να πω ότι σήμερα η μέρα είναι καλή για τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο. Είναι η πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια που μπορούμε να υποχρεώσουμε τις τράπεζες στο, ε, στα ίδια κεφάλαια που θα συμβάλλουν, δηλαδή τα ποσά τα οποία θα γράφουν στους ισολογισμούς τους να τους ανήκουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό αφορά όχι τη μία-δύο μεγάλες τράπεζες που καλύπτει η νομοθεσία της Βασιλείας, αλλά όλες τις τράπεζες της Ευρώπης. Είναι πολύ πιο αυστηρές στις προδιαγραφές για τα ίδια κεφάλαια που θα πρέπει να πληρούν οι τράπεζες όπως λέμε εμείς και έτσι ελπίζω ότι πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα άλλα κράτη θα δεσμευθούν αντίστοιχα και θα αναλάβουν τις υποχρεώσεις. Λέμε ταυτόχρονα ότι δεν θέλουμε ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως να ε, απολευστούν οι δυνατότητες για ε, πιστώσεις, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκείνες οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίες, εργασίας αυτές οι οποίες προωθούν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα στην Ευρώπη. Για αυτές λοιπόν πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα της πίστοσης και δεν θέλουμε και να λησμονήσουμε και τις κοινοτικέ πιστώσεις ε, οι οποίες μπορούν να ε, χορηγούνται χωρίς προσφορά ιδιών κεφαλαίων με εγγύηση και αυτό θα ενισχύσει βέβαια τους Δήμους και τις κοινότητες της Ευρώπης στις παραγωγικές τους δραστηριότητες. Ευχαριστώ πολύ. Στο CarSTI τώρα λέει ο Πρόεδρος. Θα σας παρακαλέσω να δείξετε και εσείς κατανόηση για το γεγονός ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε περισσότερες ομιλίες από πέντε. Η κυρία Αντζελίλη είναι η πρώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρώπη θα έχει νέους κανόνες για να ενισχύσει το τραπεζικό της σύστημα, στόχος η αποφυγή μελλοντικών κρίσεων και ε, κερδοσκοπία, αλλά και διαφάνεια επί των κερδών των τραπεζών, επί των φόρων που πληρώνουν και των ε, ε ενισχύσεων που λαμβάνουν. Όλα αυτά είναι προφορίες που θα πρέπει να καταστούν δημόσιες και να υπάρχουν σαφή όρια για τα super bonus αλλά ειδικά νέους κανόνες που θα αφορούν στην πραγματική οικονομία. Έγινε δεκτό το αίτημα, η έκκληση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ζητούσαν εγγυήσεις για την πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Πράγματι εισήχθε το, λεγόμενο support factor για τις ε, πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις για τα δάνεια. Ένα βήμα θετικό στην υπηρεσία της πραγματική οικονομίας, της ανάπτυξης και της εργασίας. Μέσα απαραίτητα προκειμένου να ενισχύσουμε την ανάκαμψη. Ευχαριστώ τον εισηγητή ε, ειλικρινά για την εξαιρετική εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αντζελίλη. Κυρία Μπρέντα το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Συμφωνία Συμβουλίου Κοινοβουλίου για τον περιορισμό των πόνους των τραπεζιτών είναι κάτι το πολύ ε, θετικό έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, συμπεριφορές κινδύνου ε, οι οποίες προωθούνται σε σχέση με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις με βάση την Βασιλεία Δυστυχώ δυστυχώς υπάρχει αντίσταση και λόμπινγκ από τον τραπεζικό τομέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τις συμπεριφορές κινδύνου στον χρηματομισθωτικό τομέα, αλλά θα πρέπει να εποπτεύουμε τους συστημικούς κινδύνους, ιδιαίτερα ως προς το shadow banking. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της ευελιξίας και των λιανικών παροχών προς τις ΜΜΕ έτσι ώστε να μην υπάρχει ψηλό κόστος για αυτή τη δανειοδότηση. Ευχαριστώ κύριε, πολύ την κυρία Πρέντεκαστ. Κυρία Σφίμπορν έχει το λόγο. Οι, συστημικές, ε, οι συστημικοί κίνδυνοι των τραπεζών αποτελούν ε, παγκόσμια πρόκληση, γι' αυτό η Επιτροπή της Βασιλείας μιλά για το μέλλον των τραπεζών ε, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κίνδυνοι. Θα πρέπει να δούμε τους μεγάλους χρηματοοικονομικούς κολοσσούς, ε, τους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πιστεύω ότι το ΟΚΑ4 θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τους μεγάλους χρηματοοικονομικούς κολοσσούς και στους συστημικούς κινδύνους των μεγάλων πιστοτικών ιδρυμάτων. Θεωρώ ότι ε, για, τις μη, για τους μη χρηματοοικονομικούς κολοσσούς ε, θα πρέπει να υπάρχουν παρόμοια μέτρα και αυτό αφορά και τα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σπίνμπεν. Νίτρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε οι πρώτοι στους G20 που εφαρμόζουμε τις διατάξεις της Βασιλείας 3 και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Θα ήθελα να τονίσω άλλο ένα σημαντικό παράγοντα. Υπάρχουν δεσμευτικά πρότυπα και ε, λαμβάνουμε όμως υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και δεν αποκλείουμε την ευελιξία μέσα στα πλαίσια της συνολικής αυτής ρύθμισης. Υπό τον πρώτο λοιπόν πυλώνα θα είναι δυνατόν να ρυθμίσουμε ε, μεμονωμένα τους αντικυκλικούς αναστολής. Επίσης, ε, καλωσορίζω και τις διατάξεις του δεύτερου πυλώνα. Τέλος, Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλίβα παρακαλώ για να ολοκληρωθεί το καρστιάρι. Κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές από την ε, συζήτηση ότι εξασφαλίστηκε μια μεγάλη επιτυχία προς την εποπτεία των ε, τραπεζών. Ε, απεδείχθη ανεπαρκής η εταιρική διακυβέρνηση όπως είχε μέχρι τώρα και έτσι οι τραπεζές εκτέθηκαν, ε, εξετέθησαν σε, μεγάλες, σε μεγάλα ανοίγματα και χρειάστηκε να καλέσουν ε, τον φορολογούμενο στη διάθεσή τους. Τώρα λοιπόν ε, βλέπουμε ότι έχουμε πάρει στα σοβαρά το ζήτημα αυτό. Ασκείται πίεση στις τράπεζες ώστε να προσφέρουν τη χρηματοδότηση τους στην πραγματική οικονομία, να επιτελέσουν δηλαδή το ουσιαστικό τους έργο. Και ιδιαίτερως θα ήθελα να χαιρετήσω τη ρύθμιση για τις ε, ρυθμίσεις των, για τα μπόνους των ε, τραπεζιτών με περιορισμό του κινδύνου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα είναι διαθέσιμα και περισσότερα κονδύλια για τη δημιουργία θέσεων και, και για να ξεφύγουμε από αυτήν την κρίση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κλέβα. Ολοκληρώνεται η συζήτηση και παρακαλώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο να έχουν το λόγο. Ο κύριος Μπαρνιέ πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να εκφράσω την ικανοποίησή μου που το σύνολο σχεδόν των βουλευτών που έλαβαν το λόγο ε, στήριξαν ε, το πνεύμα αλλά και το περιεχόμενο αυτής της πρότασης που είναι ένα θεμελιώδες κείμενο σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα προκειμένου να συναγάγουμε τα συμπεράσματα από την κρίση. Και μια που μιλάω για ευχαριστίες, να αναφερθώ σε όλους τους ε, συνεργάτες σας, ε, τους δικούς σας, τους δικούς μας, ε, διότι το θέμα είναι ιδιαίτερα τεχνικής φύσης και απέτησε μεγάλη τεχνική εμπειρία. Θα ήθελα λακωνικά να διαβεβαιώσω τον κύριο Μάλκομ και τον κύριο Τίσεν ε, και την κύριο την αποφασιστικότητα της Κομισιόν ώστε να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία που ε, συναποτελούν αυτό που λέμε τραπεζική ένωση. Πολλά που αυτά υπάρχουν, η υποπτία της ε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το κείμενο περιψηφίσματος βρίσκεται των βιών σας και με τον αυτό ο βολονταρισμό θα υποβάλουμε πριν από το θέρος ε, την πρόταση ψηφίσματος ε, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, διότι θεωρούμε ότι από νομική σκοπιά είναι δυνατόν να στηριχθούμε στην ε, υφιστάμενη συνθήκη και αργότερα όπως είπαν και οι Υπουργοί στο Δουβλίνο, μια τροποποίηση στοχευμένη ε, ίσως και στην, ε, στο της Κομισιόν το υπόδειγμα που, που βάλαμε τον Σεπτέμβριο μια μελλοντική εξέλιξη έτσι, τους συνθήκες θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω όλα τα τραπεζικά στοιχεία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε να προοδεύσουμε επί όλων των ζητημάτων ε, που, τα οποία εμπίπτουν στην ε, θέμα της εποπτείας και περιέχονται στην συνθήκη ο κ. Μπούσμαν είπε ότι το Κοινοβούλιο κάνει τι κατάλληλε προτάσεις. Να πω επίσης στον ίδιο αλλά και την κυρία Μοργάντη ότι θα παρουσιάσουμε την ε, έκθεση σχετικά με τη συνέχεια της έκθεσης Lee πριν από το θέρος, λάμβανε υπόψη όλες τις μελέτε αντικτύπου που έχουμε κάνει επί όλων των επιλογών για να δουλέψουμε αποτελεσματικά. Η Σάρων αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ε, αποδοχές και στις μπόνους. Ε, Επιβεβαιώνω ότι θέλουμε να ενισχύσουμε συστηματικά την ευθύνη των ε, μετόχων για όλες τις επιχειρήσεις και θα υποβάλουμε ένα σχετικό κείμενο. Ευχαριστώ τον κύριο Λάμπερτ και τον κύριο Κνούτ για την μαρτυρία τους. Ναι, ρυθμίζεται το χρηματοπιστωτικό τομέα. Θα πρέπει να το τονίσουμε με την λέξη κλειδί που είναι η λέξη διαφάνεια, διότι είναι η πρώτη προϋπόθεση της ε, δημιουργίας ε, ε, ευθυνών και λογοδοσίας. Η Κομισιόν θα υποβάλει λοιπόν ένα κείμενο σχετικά με το μη χρηματοοικονομικό reporting όλων των επιχειρήσεων κυρία Βίκη Φόρτ κυρία Σουέμπερ, να πω ακόμα και αν, διαφωνούμε σε αυτό το σημείο, το κείμενο που θα εγκρίνεται σήμερα είναι σύμφωνο και σύνομο με την ε, απόφαση της Βασιλείας ε, του εφαρμόζουμε σε 8.300 τράπεζες, όχι σε 30 τράπεζες όπως στις Πολιτείες, αλλά σε 8.300 τράπεζες που χρηματοδοτούν το 95% Ευρωπαϊκή Οικονομία και 4.000 αυτέ τράπεζε, τράπεζες όπως είπε ο κ. Κνούτε όπω ο κ. Μπάλτς ε, δήλωσε είναι τράπεζε ε, που κάνουν την διαφορετικότητα. 4.000 αυτέ τράπεζε τράπεζες ε, είναι συνεργατικέ τράπεζε. Ο κ. Μπλουμ, ο οποίο έχει αποχωρήσει, του προτείνω να εγκρίνει το κείμενο το οποίο προτείναμε για την καταπολέμηση των ε, των εγκληματικών δράσεων ε, να πω στον κύριο Μπέρες ότι, και τον κύριο Πρεζάδο ότι το ισότιμος ανταγωνισμός με τους άλλους εταίρους αλλά ιδιαίτερα με τους Αμερικανούς ε, την περσμένη εβδομάδα συνάντησα τον αρμόδιο υπουργό, το G20 συνέρχεται αυτή την εβδομάδα και επί πολλών θεμάτων η εφαρμογή της Βαρυσεγγίας 3 και τα τεχνικά κείμενα για τα παράγωγα το περίφημο ζήτημα των Freud Banking Organization συνεχίζουμε μια συζήτηση ειλικρινή με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, επαναλαμβάνω επίσης τα κείμενα τα οποία βρίσκονται ενώπιόν μας πέραν των όσων ήδη είπα για το shadow banking ε, με μια ρύθμιση για τα, ε, για τα χρηματοοικονομικά ζητήματα, η ισότητα όχι μόνο μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και της ε, διαφορετικότητας ε, που απαιτείται από τις τράπεζες που προσλαμβάνουν. Θα γίνει λοιπόν ε, μια τέτοια αναφορά σε περιφορά διακυβέρνηση. Κυρία Μακάρτη, τα διδάγματα που πρέπει να συναγάγουμε θα τα λάβουμε υπόψη μας γιατί ως κύριε Κλούτο όπως είχα δεσμευθεί η προστασία των καταναλωτών και των ε, βασικών καταθέσεων το κείμενο το οποίο δημοσίευσε η Κομισιόν πέρυσι για τι μακροχρόνιες επενδύσεις και τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία ε, των οποίων έχουμε ανάγκη μπορούμε να περάσουμε από έναν κανονισμό ε, διορθωτικό θα έλεγα κατασταλτικό ακόμα κάτι το οποίο απαιτείται μετά την κρίση σε μια ρύθμιση προορατική και δυναμική. Γι' αυτό λοιπόν το κείμενο που θα εγκρίνεται σήμερα είναι ε, θεμελιώδες προκειμένου να συναγάγουμε τα συμπεράσματα του, από την κρίση και να στηρίξουμε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις που θα δώσετε σε αυτή την πράσινη βιβλία και στα 30 ερωτήματα που θέσαμε, διότι πολύ από εσά ε, ενδιαφέρονται για αυτές τις μακροχρόνιες επενδύσεις. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Μπαρνιά. Κύριε Κράιτν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, θα ήθελα καταρχήν να τονίσω τα πολύ θετικά σχόλια σε σχέση με αυτό το προσχέδιο νομοθετήματος. Καταλαβαίνω ότι πολλοί από εσάς δεν νιώθετε πολύ άνετα με αυτή την πολιτική συμφωνία, αλλά όπως είπα στα αρχικά μου σχόλια, χρειάστηκε να βρούμε μία ισορροπία μεταξύ ε, συγκρουόμενων απαιτήσεων και πραγματικότητας έτσι ώστε οι τράπεζές μας να γίνουν πιο ασφαλείς εξασφολίζοντας το γεγονό ότι θα πρέπει να υπηρετούν μια ολοένα και μεγαλύτερη οικονομία. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αποτελεί συμβιβασμό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ θετικός αυτός ο συμβιβασμός και μιλάμε για έναν ενιαίο στόχο, ότι δηλαδή η Ευρώπη θα πρέπει να αναδυθεί από την παρούσα κρίση ε, ισχυρότερη έτσι ώστε να μπορέσει να υπηρετήσει τους πολίτες της, να έχουμε καλύτερη ε, εξυγίανση και τράπεζες που να μπορούν να υπηρετούν τους πολίτες. Η κυρία Μπόλς αναφέρθηκε σε αυτό τον πολύ καλό συμβιβασμό, δηλαδή φτάσαμε σε μία ισορροπία και αυτό το υποστηρίζω και εγώ. Και μιλήσαμε για επίδοση στοιχείων και μεγαλύτερη διαφάνεια που αποτελεί ένα πολύ καλό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σήμερα θα ψηφίσετε μία τροπολογία στο άρθρο 416, παράγραφος 5 Δέλτα σε σχέση με την αντιμετώπιση των ρέπος για να υπολογιστεί η αναλογία της μόχλευσης θεωρήθηκε ότι το παρόν προσχέδιο δεν είναι η σωστότερη λύση και θα πρέπει να δούμε ποια θα ήταν μια καλύτερη αντιμετώπιση, όπως είπε και η Επιτροπή της Βασιλείας. Το Συμβούλιο μπορεί να υποστηρίξει αυτή την τροπολογία μέσα στα πλαίσια του συνολικού σχεδίου και χαίρομαι που μπορώ να σας ε, το πω αυτό. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω όλους εν κατακλείδη και ιδιαίτερα τον εισηγητή για την επικοδομητική προσέγγιση, ιδιαίτερα του Κοινοβουλίου, στις διαπραγματεύσεις. Αναμένουμε τη θέση σε ισχύ του κειμένου το ταχύτερο δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κρέιτν και για να ολοκληρωθεί η συζήτηση ο κύριος Κάρας δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η συζήτηση ξεκαθαρά έδειξε σήμερα ότι η αποφασιστικότητα που είναι ορατή, αισθητή στο Κοινοβούλιο και η αίσθηση ευθύνης υλοποιούνται μέσα από τα από τις αποφάσεις αυτές. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Κάναμε μια πολύ καλή δουλειά μαζί. Θα υποστηρίξουμε την τροπολογία μετά τη συζήτηση και τη δεύτερη φράση στο άρθρο 216 θα τη διαγράψουμε. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω επιπλέον ότι η συζήτηση αυτή αποδεικνύει ότι πρέπει να πατήσουμε ακόμη περισσότερο τον γκάζι, να, να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο τους ρυθμούς για την Τραπεζική Ένωση, για την υλοποίηση της Φορολογικής Ένωσης, για την καταπολέμηση των ε, σκιωδών τραπεζών, του συστήματος των σκιωδών τραπεζών και των υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων. Και πρέπει να αλλάξουμε πλέον νοοτροπίες, πρέπει να αναλογιστούμε ότι επιβαρύνονται από το... οι διαπραγματεύσεις από το γεγονό ότι άλλαξαν τρει προεδρίε από πλευρά του Συμβουλίου στη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο, μέθοδο εργασία. Εμεί καταφέρνουμε τώρα να θέσουμε σε ισχύ από 1η Πρώτου του 2014 μια νομοθεσία υποδειγματική για ολόκληρη την ανθρωπότητα, για ολόκληρο τον κόσμο. Δεν ε, πρέπει να αφήσουμε να ε, παρακολουθεί η εφαρμογή των μετάξεων αυτών και τις νομοθεσία που θεωρούμε τόσο σημαντική. Κάτι που είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό, τα σταξιδοτικά ταμεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η αλλαγή νοοτροπία περνάει μέσα από τη διαφάνεια, τον περιορισμό των πόνου, τον περιορισμό της εκθέσεως. Η ευελιξία δεν μπορεί να αποτελέσει παράγοντα τρεύρωση του ανταγωνισμού στο βαθμό που έχουμε ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό σύστημα για τις τράπεζες και ε, αναφέρονται οι ομολογίες πρέπει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε νέε προτάσει. Ευχαριστώ πολύ. Καλύψαμε όλα τα θέματα πιστεύω και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου όσοι έλαβαν το λόγο για τα συγχαρητήρια αλλά πάνω απ' όλο του πάντε για την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάρα, Ολοκληρώνεται έτσι η κοινή συζήτηση. 12 του μεσημέρι θα γίνει ψηφοφορία σήμερα. Έχω και μία ανακοίνωση, μία πρόταση